12 τα μεσάνυχτα. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και βρίσκεται στο διαδίκτυο του στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρα της συνεδρίασης.